και αυτό δεν αποκλεί περαιτέρω συζήτηση και πιο περίπλοκο ψήφισμα να ακολουθήσει. Καλώς. Είναι ξεκάθαρη κατάσταση. Οι προτάσεις Convented και Τσίμερ είναι για μια συζήτηση τώρα και ένα ψήφισμα σε αυτή την Ολομένεια. Τώρα και συζήτηση και ψήφισμα. Ποιο είναι υπέρ αυτή τη πρότασης. Παρακαλώ με τα χέρια να σηκώσετε τα χέρια για να δούμε. Ποιοι είναι κατά. Ποιο απέχει. Νομίζω ότι εγκρίνεται η πρόταση. Τότε ε, ορίζω τις ακόλουθες προθεσμίες. Ε, η Τετάρτη στις 8, ε, Τρίτη στις 8 για τις τρο, ε, τροπολογίες την Τετάρτη στις 12 και το κοινό ψήφισμα την ε, Τετάρτη στις ε, 1 και την ε, Πέμπτη στις 12 θα γίνει η ψηφοφορία. Οπότε ορίσαμε το σχέδιο εργασίας, οπότε ερχόμαστε στην έκθεση του συναδέλφου Τσβίφκα για τη διεθνή δικαιοδοσία, αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Το λόγο έχει ο κύριος Ταντέους Τσβίφκα για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ήδη από τις αρχές των εργασιών μας ε, σχετικά με την αναθεώρηση της οδηγίας ε, περί διεθνούς δικαιοδοσίας Ένα λεπτάκι υπάρχει ένα πρόβλημα. Θα μπορούσατε να αποχωρήσετε παρακαλώ. Εκάθαρα να σας το πω. Λίγο σιγά σιγά να βγείτε και με ησυχία. Ωραία, κύριε Τσβίφκα, έχετε το λόγο. Ξεαρχίστε από την αρχή. Σας ευχαριστώ και πάλι, Πρόεδρε. Θα ήθελα λοιπόν να σας αναφέρω τα πεπραγμένα για τις εργασίες που κάναμε για την αναθεώρηση τη οδηγίας για την διεθνή δικαιοδοσία. Ήδη εξ αρχή συνειδητοποίησα πόσο περίπλοκα είναι αυτά τα ζητήματα. Η επιθυμία της ε, βελτίωσης της λειτουργία της οδηγίας αυτής που παρεπιπτόντως θεωρείται ως μια οδηγία που ε, εφαρμόζεται σωστά έδειξε τα προβλήματα και τις ανησυχίες μας. Ε, πάντως, ακόμη και για τα αμφιλεγόμενα σημεία, καταλήξαμε στις συμβαστικές λύσεις, κάναμε διάφορες συσκέψεις, ε, είχαμε έναν άτυπο τριμερή διάλογο με τις τρεις διαδοχικές ε, προεδρίες. Και νομίζω ότι μπορούμε να ελπίζουμε σε μια συμφωνία μετά την πρώτη ανάγνωση πλέον. Το πλέον σημαντικό στοιχείο ήταν η κατάργηση της εκήρυξης της εκτελεστότητας. Ε, ε, επί Προεδρίας καταλήξαμε σε μια συμφωνία βάσει βάση και των τροπολογιών που έχω συμπεριλάβει στην έκθεσή μου. Καταργείται λοιπόν η κήρυξη της εκτελεστότητας με τρόπο ώστε να βελτιωθεί η εκτέλεση εκτέλεση των αποφάσεων μειώνοντας ταυτόχρονα το γραφειοκρατικό κόστος. Ε, ταυτόχρονα θα παραμείνουν ρήτρε διασφάλισης για τους εναγόμενους ε, κάτι απαραίτητο εφόσον αποφασίζουμε την κατάργηση της κήρυξης της εκτελεστότητας καταφέραμε να καταλήξουμε σε αυτές τις συμβαστικές λύσεις διότι υπάρχει μεγάλος βαθμός εμπιστοσύνης για τα δικαστικά συστήματα των κρατών μελών. Πρόκειται για κοινή επιτυχία όλων. Στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο έχει συζητηθεί επί μακρόν ενίσχυση και η επέκταση της εφαρμογής της οδηγίας και στις τρίτες χώρες και το επωνομαζόμενο reverse effect, αντίστροφο αποτέλεσμα. Ε, στην αρχή ε, ε, ήμουν κάπως σκεπτικός γιατί το να επιφέρουμε τόσο σοβαρές αλλαγές στον κανονισμό Βρυξέλλες 1 για τους καταναλωτές, ε, παραδείγματο χάρη, με τις νέες συμφωνίες, ένας ε, πολιτής ε, που είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να προσαχθεί ενώπιον του δικαστηρίου του κράτους μέλους όπου διαμένει ο καταναλωτής. Θεωρούν όμως πολλοί ότι είναι πρόωρο το να προσπαθήσουμε να επεκτείνουμε την οδηγία και σε τρίτες χώρες. Πάντως συνιστά ένα καλό βήμα και υπερασπιζόμαστε έτσι το πλέον αδύναμο μέρος. Χάρη στην αναθεώρηση ε, της οδηγίας αναθεωρήσαμε και την ε, κατάσταση της εφαρμογής αποφάσεων ήταν δύσκολο να καταλήξουμε συμβαστική λύση για τις συμφωνίες διαμεσολάβησης. Το Κοινοβούλιο πάντως συμφώνησε ότι η ευχερέστερη και απλούστερη λύση θα ήταν να διατηρηθεί η καθιστική ατάξη για την διαμεσολάβηση, να παραμείνει εκτός του πεδίου εφαρμογής οδηγίας λοιπόν η διαμεσολάβηση, αυτό αποφάσισε το Κοινοβούλιο και αυτό πηχείται στην συμβαστική λύση στην οποία καταλήξαμε. Θα διατηρηθούν τα πράγματα ως έχουν και θα εξηγήσουμε στην αιτιολογική σκέψη τη λειτουργία αυτού του κανόνα. Θα ήθελα επίσης να αναφέρω ότι στην αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής ε, είχαμε συμπεριλάβει αυτές τις νομικές πράξεις ε, τις πράξεις κατεξουσιοδότηση και τελικά η ιδανική προεδρία επανέφερε τις πράξεις κατεξουσιοδότηση στο κείμενο. Τώρα η επιλογή του δικαστηρίου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επ' αυτού την Κυπριακή Προεδρία που κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις για αυτό το ζήτημα οι οποίες θα ενσωματωθούν στα εκτιμώντας και νομίζω ότι πλέον ο κανονισμός θα είναι αρκετά συγκεκριμένος. Τέλος Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα μέρη που ανεπλάκησαν στην διαδικασία, την Επίτροπο Ρέντινγκ, τις διαδοχικές προεδρίες, Πολωνική, Δανική, Κυπριακή, τους κοιόδης εισηγητές, τους συναδέλφους από την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα ήθελα εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να δώσω το λόγο στην Επίτροπο Ρέντινγκ. Πρόεδρε, χαίρομαι πάρα πολύ που φτάνουμε στην αναθεώρηση ε, του κανονισμού Βρυξέλλε 1. Χαίρομαι που εγγράφει στην μέση διάταξη αυτή τη ολομέλεια αυτό το θέμα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλου αυτού του πολιτικού, ιδιαίτερα προσιλωμένου συγγνώμη στο στόχο του ε, και όλο το προσωπικό που μα βοήθησε. Ε, Καταρχά, να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον κύριο Σουίφκα. Εργάστηκε με εξαιρετικό τρόπο το ίδιο και η επιτροπή του. Στη συνέχεια να ευχαριστήσω τις, Πολωνι... τις τρεις προεδρίες, Πολωνική, δανική και Κυπριακή, χάρη στις οποίες με εύρυθμο τρόπο θα εξαρτηθεί στο Συμβούλιο του Δεκεμβρίου πλέον ο αναθεωρημένος κανονισμός. Ε, συνιστά αυτό μεγάλη επιτυχία για τους πολίτες, για τις επιχειρήσεις, καθώς και για την ενιαία αγορά. Και πρόκειται για μία από αυτές τις επιτυχημένες ε, ε, ιστορίες ε, που δημιουργούν έναν ευρωπαϊκό χώρο δικαιοσύνης και που καταδεικνύουν ότι η δικαιοσύνη μπορεί να τονώσει και την ανάπτυξη. Εδώ μιλάμε για 500 εκατομμύρια καταναλώτες, κυρίως για μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν πλήρω το δυναμικό τη εσωτερική αγορά λόγω ε, εσωτερικών φραγμών. 40% των επιχειρήσεων ε, θα ε, επεκτείνουν τι διασυνοριακέ συναλλαγέ του κατά πάσα πιθανότητα δηλώνουν αν απλουστευθούν οι διαδικασίε για την επίλυση των δικαστικών διαφορών. Ακριβώ αυτό κάνουμε τώρα. Έρουμε τα γραφειοκρατικά εμπόδια που συνεπάγονται επιπρόσθετο κόστο και νομική ανασφάλεια για του συμβαλόμενου. Ε, και αυτό υπηρετεί το στόχο μας, ε, δηλαδή ε, την δημιουργία μέσω εσωτερικής αγοράς που θα είναι ελκυστική για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Με την αναθεώρηση του κανονισμού Βρυξέλλες 1 κάνουμε μια σημαντική συνεισφορά, όπως σωστά είπε ο συγγητή, Καταργούμε την διαδικασία κήρυξης εκτελεστότητας των αποφάσεων. Πρόκειται για μια διαδικασία που στις περισσότερες περιπτώσεις δεν είναι αναγκαία, αλλά κοστίσει 2.000 ευρώ ανά υπόθεση για τις διατυπώσεις. Ε, μελλοντικά θα καταργήσουμε αυτή τη γραφειοκρατία και το όφελος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα είναι 47 εκατομμύρια το χρόνο. Θα κάνουμε αυτό που κάνει το Ηνωμένο Βασίλειο εδώ και πάρα πολύ καιρό για το άρθρο 4 δηλαδή του συντάγματος όπου αναφέρεται η αρχή της αξιοπιστίας της εσωτερικής αγοράς. Αυτό θα το επιτύχουμε με την κατάρριση εκτελεστότητας. Στη συνέχεια, επιλογή του δικαστηρίου. Η συντριπτική πλειοψηφία των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων περίπου 40% των επιχειρήσεων και 90% των μεγάλων επιχειρήσεων χρησιμοποιούν αυτή την επιλογή των συμφωνιών παρέκτασης της δικαιοδοσίας. Ε, ε, η αναθεώρηση που είναι τώρα επιτάπητος μας προσφέρει την απαιτούμενη νομική ασφάλεια για να το επιτύχουμε αυτό. Στη συνέχεια έχουμε και τις εξωτερικές διαστάσεις του κανονισμού Βρυξέλλες 1 όταν ε, δηλαδή υπάρχουν δίκες όπου εμπλέκονται τρίτες χώρες για την υπεράσπιση του αδύναμου μέρους μεριμνήσαμε το ώστε όλοι ε, φυσικά και νομικά πρόσωπα στην Ευρώπη θα έχουν πρόσβαση στη δικαιοσύνη ανεξαρτήτως τόπου διαμονής. Πρόκειται για ένα πάρα πολύ απτό όφελος ε, για τους Ευρωπαίους πολίτες. Τέλος υπάρχει και το ε, δύσκολο θέμα της διαμεσολάβησης. Κύριε Τσβίφκα θα δεχτούμε αυτήν την συμβαστική λύση που κατά τη γνώμη μου συνιστά ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση Πρόεδρε. Θα έλεγα ότι πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα προς ένα ουσιαστικό ευρωπαϊκό χώρο δικαιοσύνης και θα ήθελα να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο για την υποστήριξη που μας προσφέρει. Θα υπεραμεινθώ της πρότασης του Κοινοβουλίου ενώπιον του Συμβουλίου και το Δεκέμβριο θα ήθελα να γιορτάσουμε την κοινή μας επιτυχία. Ευχαριστούμε την κυρία Επίτροπο. Τώρα από την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, η κυρία Ρέγκνερ ε, θα μας δώσει τη θέση της Επιτροπής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμη Επίτροπε Ντίνκ, θα ήθελα καταρχάς μετά από δύο χρόνια διαπραγματεύσεων να ευχαριστήσω τον ε, κύριο Τσβίφκα για την επιμονή του και για την ε, τρόπο που διεξήγαγε τις διαπραγματεύσεις και τις ε, προεδρίες, την Κυπριακή που είναι τώρα και την Πολωνική και την Δανική που επικοδομητικά συνεργάστηκαν. Ε, πρόκειται για μια επανάσταση. Εμείς ως νομοθέτες ε, έχουμε καταφέρει να βελτιώσουμε μια νομοθεσία για τους εργαζόμενους και τους καταναλωτές ο κανονισμός ε, για τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις ε, θα αναθεωρηθεί έτσι ώστε να ε, συμπληρώσει μια πολύ καλά λειτουργούσα νομοθεσία στην εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό ειδικά για την ομάδα των σοσιαλδημοκρατών που εκπροσωπώ. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις ε, η κατάργηση της διαδικασίας κήρυξης εκτελεστότητας είναι μια βασική διαδικασία ε, που παρά τις αμφιβολίες κατάφερε να ευοδοθεί. Ε, επίσης, με τον κανονισμό για τα τρίτα κράτη ε, δεν καταφέραμε ε, να κάνουμε αυτό που θέλαμε, αλλά τουλάχιστον μπορέσαμε να ασχοληθούμε με ατομικές υποθέσεις ε, για την προστασία του αδυνάμου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό οι διαπραγματεύσεις για αυτόν τον κανονισμό. Έχουν να κάνουν και με την Πράσινη Βίβλο 2009, στην έναρξη δηλαδή της νομοθετικής περίοδου. Δύο χρόνια διήρκησε η αναδιατύπωση. Είναι ε, πολύ ιδιαίτερη αυτή η περίπτωση. Είναι μια ρικάστα αυτή η αναθεώρηση. Κατά την άποψή μου αυτή ε, η διαδικασία είναι μια απλό, απλούστευση για επιτάχυνση των διαδικασιών. Η Βρυξέλλες 1 δεν είναι ένα θέμα διαμφισβήτητο ε, όπως είναι συνήθως για αυτές τις διαδικασίες και γι' αυτό η διαδικασία δεν ήταν καθόλου σύντομη. Ε, γιατί ήθελε λοιπόν η Κομισιόν να υπάρχει αυτό το recast. Ε, από την άποψή μου, ε, δημοκρατικά αυτό είναι λυπηρό. Και η διαθεσμική συμφωνία με την Κομισιόν πρέπει να τύχει επεξεργασίας. Δεν πρέπει ε, η εκτελεστική εξουσία να περιορίζει την νομοθετική με αυτόν τον τρόπο, να προτείνονται αλλαγέ φυσικά. Το σημαντικό είναι να τελειώσει αυτή η διαδικασία. Προτείνω λοιπόν για το μέλλον, για την ε, Σύμβαση Βρυξέλλες 1, να υπάρχει και ένα θέμα για τις ε, κινητοποιήσεις ε, τις εργασιακές έτσι ώστε να υπάρχει μια συνοχή με τα ουσιαστικά ε, δικαιώματα. Πρέπει να δούμε ποια είναι τα δικαιώματα τα οποία θα πρέπει να αποζημιώνονται. Αυτό προβλέπει ότι ε, όταν μιλάμε για απεργίες θα πρέπει να εφαρμόζεται το δίκαιο της περιοχής όπου γίνεται η απεργία. Αυτό πρέπει να το προσέξει η Κομισιόν ε, και εμείς στο Κοινοβούλιο προσέχουμε πάρα πολύ αυτό το σημείο. Ευχαριστούμε τη συνάδελφε. Ε, δέχεστε την μπλε κάρτα του κυρίου Στογιάννου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Ρέτνερ, είπατε κάνα δύο φορές ότι μιλάτε υπό την ιδιότητα του σοσιαλδημοκράτη. Παρουσιάσατε την θέση της ομάδας σας. Έπρεπε να εκφράσετε όμως την θέση της ε, ε, Επιτροπής Απασχόλησης. Είχατε τρία λεπτά στη διαθέσή σας και μιλήσατε για την γνωμοδότηση αυτής της Επιτροπής μόνο στα τελευταία 30 δευτερόλεπτα της παρέμβασής σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ευκαιρία αυτή να μου δώσετε μια απάντηση ούτω ώστε να μπορείτε να δώσετε περισσότερε λεπτομέρειες όσον αφορά τη θέση της Επιτροπής σας. Κύριε κύριε Στογιάννοφ. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει αυτός ο ενθουσιασμός από τα μέλη. Ε, το είπα μία φορά μόνο ότι ανήκω στους Σελδημοκράτες, είμαι περήφανη γι' αυτό. Ε, θεωρώ ότι η θέση της Επιτροπής Απασχόλησης έχει να κάνει με τις εργασιακές κινητοποίησεις και το ε, έθεσα αυτό το θέμα. Αυτή την ε, πρόταση λοιπόν ε, σας την θέτω προς αμφισβήτηση αν θέλετε. Ε, τώρα δίνω το λόγο στον κύριο Μπελτασάρη. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί επίτροπες, συνάδελφοι. Τώρα, αυτή την εποχή μιλάμε για μεγαλύτερη ε, ολοκλήρωση. Για κάποιους εθνικιστές ε, νοσταλγού αυτό σαν πρόκληση και θε, καλούμαστε να ψηφίσουμε αναθεώρηση ενό κανονισμού που αποτελεί τη βάση τη δύσκολη διαδικασία, αλλά απαραίτητη τη διαδικασία εναρμόνιση και ε, εναρμόνιση των διαφόρων νομικών συστημάτων κρατών μελών. Επιτρέψτε μου να συγχαρώ τον συνάδελφο Ζέτερ για τη δουλειά την περίφημη που έκανε και μετά από δύο χρόνια δύσκολων διαπραγματεύσεων ο κ. Ζεύκα κλείνει αυτή η διαδικασία αναθεώρηση των κανονισμού που είναι θεμελιώδη για του ε, πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Βρυξέλλε 1 συμπεριλαμβάνει σημαντικότητε διατάξει για να υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης δικαιοσύνη με αντιμετώπιση από τα αρμόδια δικαστήρια εντός της Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί καθορίζονται κοινέ διατάξεις σε θέματα αστικά και εμπορικά και διευκρινίζει ποια είναι τα αρμόδια δικαστήρια σε μια διαφορά δυσυνοριακή και καθιστά εκτελεστές τις διάφορες ε, ποινές των διαφόρων κρατών μελών. Χρειάζονται προσαρμογή στον κανονισμό για να δοθεί συνέχεια στη βούληση που υπάρχει να δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό χώρο δικαιοσύνη που προωθεί την ασφάλεια δικαίου και την προβλεψιμότητα των αποφάσεων, διευκολύνοντα έτσι τι υπερεθνικέ ε, συναλλαγέ και ενισχύοντα την ενιαία αγορά. Εγώ πιστεύω ότι η πρόοδος προς μια βαθύτερη εναρμόνιση των διαφόρων διατάξεων του αστικού δικαίου θα πρέπει να προχωρήσουν με προσοχή, συνετά, ούτω ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια δικαίου και η προστασία των ε, λιγότερο ισχυρών μερών. Γι' αυτό τον λόγο συμφωνώ με την προσέγγιση που διαθέτησε ο εισηγητής υπέρ του καταναλωτού οι οποίοι θα ευνοηθούν από την αρχή της προστασίας ε, του πλέον αδυνάμου. Είναι μια αρχή βάση της οποίας σε μια νομική διαφορά μεταξύ καταναλωτού και επιχείρησης ο καταναλωτής θα μπορεί πάντα να επιλέξει να στραφεί προς μια ε, στη δικαιοσύνη του κράτους μέλους στο οποίο ε, κατοικεί. Αναλόγως συμφωνώ με την συνετή προσέγγιση του συναδέλφου ε, Ζήφκη όσον αφορά την εκτελεστότητα. Κατάργηση αυτή θα επιταχύνει ακόμα πιο, ε, την αναγνώριση των κυρώσεων και αν χρειάζεται θα πρέπει να διατηρηθούν ε, ρήτε διαφύλαξης διαφύλαξη την προστασία των δικαιωμάτων των διαδίκων. Μπορεί να υπάρχει δυνατότητα αμφισβήτηση προσβολής κάποιε αποφάσεις αν θεωρούν, θεωρούν ότι το δίκαιό του έχει παραβιαστεί και αν η απόφαση είναι αντίθετη με τη δημόσια τάξη του κράτους αναφοράς. Ξανά θέλω να συγχαρώ τον εισηγητή και τους σκιώδεις εισηγητές για αυτή την προσπάθεια. Ελπίζω ότι θα πετύχουμε ευρεία συνένεση διοργανική πολιτική επί του κανονισμού που αποτελεί τη βάση για τη δικαστική και πολιτική συνεργασία και δείχνει αποφασιστικότητα πολιτική όσον αφορά την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε συνάδελφε. Μασίπ Ιντάλγκο, επόμενος. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο κύριο Χιντάλγκο. Πρόεδρε, εκείνοι που έχουν επαγγελματική εμπειρία ή εκείνοι που έχουν υποφέρει από τις διάφορες δικαστικές διαδικασίες λόγω αργών διαδικασιών, όλοι αυτοί θα εκτιμούν τις κινήσεις που κάνουμε για την κατάργηση της εκτελεστότητας και την προσπάθεια προσέγγισης των νομοθεσιών. Είναι ένα ακόμα βήμα που γίνεται βήμα το οποίο θα οδηγήσει σε ολοκλήρωση κάτι το οποίο καθημερινά προσπαθούμε να πετύχουμε. Και αυτό είναι και ο λόγο ύπαρξη άλλωστε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πριν από 8 χρόνια ήμουν στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων και συζήτησα το θέμα με δύο υπουργού τη Ολλανδική τότε Προεδρία. Συζητήσαμε το συγκεκριμένο θέμα το οποίο ε, οδήγησε σε κάποια αποτελέσματα και καρποφόρησε. Και συγχαίρω γι' αυτό τον κύριο Ζεύκα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όλες τις προεδρίες οι οποίες κατέβαλαν προσπάθειες έκτοτε. Πιο συγκεκριμένα την Ισπανική Προεδρία, θέλω να ευχαριστήσω, τον κύριο Καμπάνιο και τον Χουάν Κάρλος Κάμπος, τον Υπουργό και το Γενικό Διευθυντή μεταξύ άλλων τη αρμόδια υπηρεσία. Σα ευχαριστώ όλου για την προσπάθεια. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Λίχτεμπεργκερ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ καταρχάς ε, τον εισηγητή και τους συναδέλφους και τις συναδέλφισες που για δύο χρόνια από κοινού με αφοσίωση εργάστηκαν κάθε φορά που υπήρχε μια συνάντηση με το Συμβούλιο και υπήρχαν όλες οι αντιστάσεις, υπήρχε αμφιβολία, όμως τελικά ε, καταφέραμε να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Η διασυνοριακή, το διασυνοριακό εμπόριο ε, πάνω απ' όλα στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται κανόνες για τα πράγματα αυτά που ε, πρέπει να είναι τόσο ξεκάθαρα ώστε οι αδύναμοι να μην βρίσκονται σε δύσκολη θέση. Αυτό σημαίνει ότι αυτό που κάναμε εμείς ε, σε αυτό τον κανονισμό ήταν η προσπάθεια ε, πρώτον να δώσουμε πρόσβαση στο δίκαιο, ε, να είναι κατανοητό το δίκαιο και να είναι ξεκάθαρο. Να βελτιώσουμε αυτά τα στιγμία. Σημαντικό είναι η αμοιβαία αναγνώριση. Θεωρώ ότι ε, τα κράτη-μέλη που εκπροσωπούνται σε αυτό το σώμα, τα 27 κράτη-μέλη, θεωρούν το καθένα ότι το δικό του σύστημα είναι, νομικό σύστημα είναι το καλύτερο στον κόσμο. Όμω, όταν συνεργαζόμαστε και θέλουμε να συνεργαστούμε, πρέπει να μαθαίνουμε ένα από τον άλλον και να ε, μάθουμε να αναγνωρίζουμε τις αποφάσεις ο του άλλου. Αυτό πάντοτε ε, πισκιαζόταν από μεγάλη δυσπιστία. Φυσικά ο καθένας θέλει σε κάθε περίπτωση να μπορεί να βρει ένα παράδειγμα όπου το δικό του δίκαιο είναι καλύτερο από ένα άλλο. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι αυτή η αρχή είναι πανταχού παρούσα. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό βήμα ε, το ότι μπορέσαμε να ενισχύσουμε τη θέση του αδυνάμου και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους καταναλωτές και τις καταναλώτριες ε, που κάνουν διασυνοριακές συναλλαγές να έχουν νέες ευκαιρίες πλέον στα χέρια τους ώστε πιο γρήγορα, πιο καλά και πιο ξεκάθαρα να ε, εποφελούνται από τα δικαιώματά τους. Ε, χαίρομαι επίσης και για τη ρήτρα αναθεώρησης. Ε, πραγματικά θα χρησιμοποιήσουμε αυτό το θέμα, αλλά όπως ε, υπόθηκε αυτό έχει να κάνει με τη ρήτρα αναθεώρησης. Σήμερα αυτό που αποφασίζεται είναι ένα σημαντικό βήμα, αλλά δεν είναι το τελευταίο. Θα μας βοηθήσει όμως να δώσουμε ε, την δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους πολίτες που, και να, να γίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση πιο ξεκάθαρη για αυτούς. Ε, ο κύριος Πάσχα Γιάροσλαφ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κύριε Επιτροπέ. Ε, εκτιμώ ιδιαίτερα τις προσπάθειες της Κομισιόν μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δημιουργήσει σωστούς μηχανισμούς. Θεωρώ ότι η λύση ε, του προβλήματος ε, δεν κινείται όμως στη σωστή κατεύθυνση. Τα νομικά συστήματα των κρατών μελών εδώ και εκατοντάδες χρόνια έχουν ε, υποστεί διάφορες εξελίσεις με βάση τις δικές τους κουλτούρες και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες. Έτσι λοιπόν είναι διαφορετικό το δίκαιο σε κάθε χώρα. Ας πούμε στην Ισπανία ε, πολλές φορές ε, ε, έχουμε ανθρώπους που ζητούν να πάρουν το παιδί από τη μητέρα που ζει σε μια άλλη χώρα ή στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μπορεί να γίνει ταυτόχρονα κάτι παρόμοιο σε οικογένειες που έρχονται στην Ηνωμένο Βασίλειο για να βρουν δουλειά. Θεωρώ λοιπόν ότι τέτοιες αποφάσεις δεν είναι σωστές. Έτσι λοιπόν, πρέπει να είμαστε πάντα μέσα στα πλαίσια της πραγματικότητας. Έτσι λοιπόν όσον αφορά την εκτέλεση στο εξωτερικό μιας απόφασης ε, θα πρέπει να υπάρχει το δικαίωμα προσφυγής ε, κατά αυτής της εκτέλεσης. Ο κύριος Τσιβίφκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Πάσκα, δεν συμφωνείτε ότι θα ήταν πολύ πιο λογικό και πολύ πιο πρακτικό και πιο αποτελεσματικό αν η πολιτική σας ομάδα συμμετείχε στη δουλειά που έγινε επί του θέματος κατά τη διάρκεια όλης της περίοδου που επεξεργαζόμασταν τις Βρυξέλλες 1 παρά να προβαίνετε σε τις δηλώσεις στην Ολομέλεια πολιτικές δηλώσεις που δεν έχουν μεγάλη σχέση με το συγκεκριμένο θέμα και την εργασία που κάναμε. Αγαπητέ συνάδελφοι. E, Ευχαριστώ. Εγώ προσωπικά δεν είμαι στην Επιτροπή σας. Είμαι στην Ήτρε. Και γι' αυτό δεν συμμετείχα καθόλου σε αυτή την εργασία. Όμως ε, συμμετέχω ε, στην ανταλλαγή απόψεων και αν θέλετε να δεχτείτε την άποψή μου, τότε μπορούμε να συνεργαστούμε πολύ καλά. Ευχαριστώ. Τον λόγο ο κύριος Χένα. Ευχαριστώ. Διαπιστώνει κανεί στην πράξη ότι λειτουργεί ο Ευρωπαϊκό χώρο ει βάρο των πολιτών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αντίθετα, είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τι μεγάλε επιχειρήσει και για του πολίτε που μπορούν να πληρώνουν σειρέ δικηγόρων στη χώρα του και σε διεθνέ επίπεδο. Ε, και με χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι με υπόθεση που εμπλέκει τη Γαλλία και την Ισπανία ε, και απασχολεί τον τύπο αυτή τη στιγμή. Με τη νέα πρόταση προτείνεται επιδείνωση της κατάσταση και έτσι μια απόφαση που έχει εκδοθεί σε ένα κράτος μέλος κηρύσσεται εκτελεστή χωρίς καμία ενδιάμεση διαδικασία σε ένα άλλο κράτος και έτσι αμφισβητείται το δικαίωμα ε, της αμφισβήτησης ε, της απόφασης ενός ε, κράτους μέλους με την επίκληση παραδείγματος χάρη της μη συμμόρφωσης με τις αρχές περιδημοσίας τάξη ενός κράτους μέλους. Πρόκειται για οπισθοδρόμηση. Ε, δεν επανεξετάζεται το θέμα της αρμοδιότητας ε, του δικαστηρίου βάσει της νέας πρότασης και θα λειτουργεί σαν ένα, ένα αυτόματος μηχανισμός ε, πλέον το καινούριο σύστημα και με την υπόθεση Ωρέρ Μαρτά νομίζω βλέπουμε ότι πρόκειται για ένα, μια αυταρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης πέρα από την ελεύθερη και καταστροφική οικονομική πολιτική πολιτική. Ευχαριστώ. Τελευταίος. Εκ μέρους των ε, ομάδων, ο κύριος Στοβιάνο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα συνεχίσω πάνω σε αυτά που έλεγε ο κύριος Σίφκα. Έχω ένα ερώτημα. Αν λειτουργεί τόσο καλά ο κανονισμός, χρειάζεται μεταρρύθμιση τώρα Έθεσα το ερώτημα και έφτασα σε δύο ανησυχητικά συμπεράσματα. Τα συνήγαγα από αυτά που είπε η κυρία Ρέντινγκ. Πρώτα απ' όλα η επιλογή του δικαστηρίου. Είπε η κυρία Ρέντινγκ ότι 90% των υποθέσεων, το, στο 90% των υποθέσεων μεγάλες εταιρείε προτιμούν μία συμφωνία για την επιλογή δικαστηρίου. Διότι μεγάλε εταιρείε ισχυροί θέλουν να επιβάλλουν ένα δικαστήριο που θεωρούν ότι είναι πιο χρήσιμο, πιο ωφέλιμο για την εταιρεία. Δεν νομίζω ότι οι μικρές εταιρείε είναι εκείνες που κερδίζουν από τον κανονισμό. Είπε η κυρία Ρέντινγκ μετά ότι αυτό μας φέρνει πιο κοντά, αυτός ο κανονισμός μας φέρνει πιο κοντά στη θέση των Ηνωμένων Πολιτειών, δηλαδή μεγαλύτερο φεντεραλισμό. Εγώ είμαι υπέρ ε, της Ευρώπης των Εθνών και συμφωνώ με αυτά που μας είπε ο κύριος Πάσκα. Αυτή η ομοσπονδοποίηση της Ευρώπης για μένα είναι κάτι απαράδεκτο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Έχουμε τρεις συναδέλφους για την ε, γενική συζήτηση. Η κυρία ε, Αγγελίλη ξεκινά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αντιπρόεδρε Ρέντινγκ. Σα συγχαίρω και σας και τον συγκητή για την ολοκλήρωση του περίπλοκου θέματος που φτάνει στο τέρμα μακράς και περίπλοκης συζήτησης. Τελικά υπάρχει μια συμφωνία με το Συμβούλιο και αντικατοπτρίζεται πλήρως η θέση του Κοινοβουλίου ξεκινώντας από την κατάργηση ε, της εκτελεστότητας άνευ εξαιρέσεων. Η εκτελεστότητα αντιπροσωπεύει ένα βήμα ιδιαίτερα σημαντικό, διότι με τέτοιες καταργήσεις Εκ των πραγμάτων καταργείται δικαστική ενδιάμεση διαδικασία που κατέδειξε στην πράξη ότι έγινε πλέον μία απλή τυπική διαδικασία και μειώνεται το κόστος και ο χρόνος επίλυσης των διασυνοριακών διαφορών. Σίγουρα θα υπάρξει μεγαλύτερη προστασία για τους πολίτες που μπορούν να στραφούν προς το δικαστήριο της χώρας καταγωγής τους για διαφορές και κατά εταιριών των οποίων οι δραστηριότητες ασκούνται και σε τρίτες χώρες. Θα υπάρξουν σίγουρα καλύτερες συμφωνίες όσον αφορά την επιλογή του αρμοδίου βήματος για να εμποδιστούν οι τακτικές ε, ανορθόδοξες διαδικασίες. Θα διευκολυνθεί έτσι περαιτέρω η ελεύθερη κυκλοφορία των αποφάσεων και πάνω απ' όλα θα υπάρξει καλύτερη πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Μικρότερη γραφειοκρατία, λιγότερες σπατάλες και χρονικές και οικονομικές. Ασφάλεια δικαίου, μεγαλύτερη προσβασιμότητα. Πιστεύω ότι σε εποχές κρίσεων οι πολίτες, οι οικογένειες και επιχειρήσεις μπορούν να εκτιμήσουν πολύ αυτή την μείωση της γραφειοκρατίας και την απλούστευση των διαδικασιών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ αγαπητή Η κυρία Παμπενόβα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε. Για το νομοθετικό πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρειαζόμαστε τέτοια μέτρα που να ε, ισχύουν διασυνοριακά. Χρειαζόμαστε κανόνες ε, οι οποίοι δεν θα αποτελούν εμπόδιο. Υπάρχουν συγκεκριμένα παραδείγματα γι' αυτό και ε, για να μην ξανασυμβούν χρειαζόμαστε κανονισμούς, κανόνες ε, που θα εμποδίζουν ε, τη σύγκρουση συμφερόνων όσον αφορά στην αναγνώριση των αποφάσεων μεταξύ των κρατών μελών. Είναι πολύ σημαντικό για τους επιχειρηματίες στην Ευρώπη να είναι επιτυχημένη η διαδικασία Βρυξέλλες 1. Χρειαζόμαστε λοιπόν συγκεκριμένες διατάξεις να τις αναδιατυπώσουμε. Υποστηρίζω λοιπόν την κατάργηση της κήρυξης εκτελεστότητας γιατί έτσι θα βελτιωθεί η διαδικασία αποφάσεων και θα βελτιωθεί έτσι ο κανονισμός ώστε να βελτιωθεί και η ασφάλεια δικαίου. Πρέπει λοιπόν να είναι προτεραιότητά μας να προστατεύσουμε περισσότερο τους αδύναμους, να τους δώσουμε δυνατότητα για μια ε, δίκαιη δίκαια και να έχουμε και μία αναφορά στις διαδικασίες των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Η κυρία Τικάου, ευχαριστώ Πρόεδρε. Σχετικά με, τη, με αυτόν τον Ευρωπαϊκό χώρο δικαιοσύνης, ένας από τους βασικούς στόχους είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη, κυρίως μέσω της αμοιβαία αναγνώρισης των δικαστικών και εξοδικαστικών διαδικασιών σε αστικές υποθέσεις. Για να εμβαθύνουμε τη συνεργασία, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εγκρίνει αποφάσεις σε σχέση με τις δικαστικές αποφάσεις με ίδια συνοριακή εφαρμογή για να παγιοποιήσει έτσι την ενιαία αγορά η αμοιβή εμπιστοσύνη ως προς τη λειτουργία των ενών συστημάτων των κρατών μελών. Είναι μια βασική αρχή. Βάσει αυτής της αρχής οι αποφάσεις που εκδίδονται σε ένα κράτος θα αναγνωρίζονται σε όλα τα υπόλοιπα χωρίς κάποια επιπρόσθετη διαδικασία. Αυτό θα μειώσει και τις προθέσεις προθεσμίες αλλά και το κόστος για όλους. Απλωστεύονται έτσι όλες οι διαδικασίες ε, και διατηρείται και διαφυλάσσεται η αυτονομία των διαδίκων. Για να λειτουργήσει αυτό το σύστημα θα πρέπει να προβλέπετε δυνατότητα διεξαγωγής δίκης ανεξαρτήτως τόπου διαμονής ε, του εναγωμένου. Τα άρθρα 19 και 20 έχουν ιδιαίτερη σημασία κατά τη γνώμη μας, κυρίως οι διαδικασίες που σχετίζονται με έναν εργαζόμενο που δεν έχει την επίσημη διαμονή του σε ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορεί όμως να κινήσει, να γύρει κάποια αγωγή εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα για την προστασία των καταναλωτών, θα υποφελείται από ιδιαίτερα ευνοϊκέ διατάξει. Όλα αυτά είναι σημαντικά βήματα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ όλους του ιδιαίτερου που αναφερθήκαμε στην Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Τώρα στη διαδικασία Κατστιάη δεν έχει ζητήσει κανείς ε, το λόγο. Υπάρχει αυθορμήτω κάποιο που θα ήθελε να πάρει το λόγο, αν όχι να δώσουμε το λόγο στην Επίτροπο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, πρόκειται όντω για μια μείζωνα μεταρρύθμιση που προωθείται από όλα τα θεσμικά όργανα και όλα τα θεσμικά όργανα πρέπει να είναι υπερήφανα για αυτήν, διότι χάρη σε αυτή την αναθεώρηση μπορούμε να ε, γεφυρώσουμε τα χάσματα ανάμεσα στα διάφορα δικαστικά ε, συστήματα των κρατών μελών. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό το βήμα παρότι δεν μπορέσαμε να καταλήξουμε συμφωνία για όλα τα ζητήματα όπως η διαμεσολάβηση ή οι κανόνες ε, περί διεθνούς δικαιοδοσίας όταν μιλάμε για προβλήματα και διαφορές στον εργασιακό χώρο. Θα ακολουθήσουν όμως και άλλα βήματα, θα συνεχιστεί η διαδικασία και θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που τόνισαν το βαθμό στον οποίο έχουμε προοδεύσει για πολλά από αυτά τα ζητήματα και χωρίς την συνθήκη της Λισαβόνας δεν θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει όλα αυτά τα απαραίτητα ε, βήματα απαραίτητα ούτως ώστε να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη οι οικονομικέ και δικαστικές διατάξεις όλων των κρατών μελών έτσι δίνουμε σάρκα και οστά στην αμοιβή αναγνώριση των δικαστικών αποφάσεων. Δηλαδή αναγνωρίζουμε αποφάσεις που έχουν εκδοθεί από εθνικά ε, δικαιοδοτικά όργανα και θεωρούμε ότι δεν υπάρχει καμία διαφορά στην εφαρμογή της απόφασης, ε, ανεξαρτήτως δηλαδή του κράτους μέλους. Ακριβώς αυτό χρειαζόμαστε αν θέλουμε να επιτύχουμε ουσιαστική ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, όχι μόνο των αγαθών και των υπηρεσιών, αλλά και των πολιτών και δικαστικών αποφάσεων που τους αφορούν. Αυτό το σχέδιο αναθεώρησης που εξετάζουμε σήμερα θα είναι ιδιαίτερα επωφελές ε, για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις και από ιστορικής πλευράς ε, θα συνιστά ένα βήμα καμπή που θα μας οδηγήσει εν τέλει στη δημιουργία ενός γνωσίου ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης. Ευχαριστώ την κυρία ε, Αντιπρόεδρο της Επιτροπής. Ο εισηγητής έχει το λόγο για το τέλος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω. Ευχαριστώ τους συναδέλφους για τη συζήτηση. Ευχαριστώ που μοιραστήκατε τις απόψεις σας ε, για το θέμα αυτό. Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που μας είπε μόλις τώρα η Επίτροπος, η κυρία Ρέντι, Να προσθέσω κάτι. Όταν ξεκινήσαμε πριν από δύο χρόνια την επεξεργασία του εγγράφου, όλοι μας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όλοι μας είχαμε το δικό μας όραμα σχετικά με το πώς θα έπρεπε να προοδεύσουν οι εργασίες και ποιο θα έπρεπε να είναι το τελικό αποτέλεσμα. Σήμερα θέλω να πω ένα πράγμα. Είμαι απόλυτα σίγουρος ότι δεν έχουμε καταστρέψει την, ε, ένα νομικό μέσο που λειτουργούσε. Καλά, αντίθετα, βελτιώσαμε τη λειτουργία του. Και ε, α, έχει ενισχυθεί ο χώρος της ε, δικαστικής συνεργασίας στην Ευρώπη. Οι πολίτες, ε, οι εργοδότες, οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων θα έχουν στα χέρια τους ένα εργαλείο που θα τους επιτρέψει να λειτουργούν καλύτερα εντός της ενιαίας αγοράς. Είμαι πεπισμένος ότι θα υιοθετήσει το έγγραφο το Κοινοβούλιο και περιμένω με ανυπομονησία να το εγκρίνει και το Συμβούλιο, τόσο ώστε όλοι να μπορούμε να πούμε ότι κάναμε καλή δουλειά. Ξανά ευχαριστώ όλους σας. Ευχαριστούμε πολύ τον ε, εισηγητή. Κλείνει λοιπόν η συζήτηση. Ε, αύριο στις 12 θα έχουμε την ψηφοφορία. Ερχόμαστε λοιπόν στο επόμενο θέμα της ημερήσια διάταξης. Πρόκειται για την προφορική ερώτηση προς την Επιτροπή.